της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκοσμίες αλυσίδες αξίας. Σας δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το παγκοσμιοποιημένο σύστημα μας στηρίζεται σε διαδικασίες παραγωγής κατακαιρματισμένες. Τα περισσότερα αγαθά είναι μια σύνθεση διαφορετικών λειτουργιών στις τέσσερις γωνιές ε, του πλανήτη μερικές φορές, ε, σε αναζήτηση εταιρικών σχέσεων, αναζήτηση υλικών, πρώτων υλών και περισσότερες φορές για το χειρότερο. Μια κοινά εργατικά, ε, φοροδιαφύγη. Όλες αυτές οι λειτουργίες ε, συντονίζονται από διεθνείς επιχειρήσεις μέσω συμβατικών εταιρισμών ή υπεργολαβιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρώτος εξαγωγέας και εισαγωγέας στον κόσμο αγαθών και υπηρεσιών μπορεί και θα λέγα πρέπει να κάνει την πολιτική της, την εμπορική, ένα μοχλό για να καταστήσει αυτές τις αλυσίδες ε, εργαλείο για την αηφόρα ανάπτυξη και να οδηγήσει σε μια πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη στιγμή ε, η διαφάνεια και η έλψη ε, ευθύνη αυξάνει τους κινδύνους εκμετάλλευσης των εργαζομένων, το μη σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων και την υποβάθμιση σε περιβαλλοντικό και σε άλλους τομείς. Αυτή η έκθεση γράφεται σε μια πολιτική όπου επικρίνεται από τους πολίτες που ζητούν μια πιο δίκαιη, πιο διαφανή παγκοσμιοποίηση. Αυτή η έκθεση απαιτεί από την Κομισιόν να ε, λάβει μια σειρά από μέτρα για να κάνει τις ε, ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξιών πιο υπεύθυνε και πιο διαφανείς. Για να, θα, μπορούσα να αναφερθώ στην συμπερίληψη στις εμπορικές συμφωνίες, ένα κεφάλαιο κατά της φοροδιαφυγής και επίσης την λήψη πρωτοβουλειών ε, για να υπάρχει επαγρύπνηση στις εταιρείες σε ένα πλαίσιο με περιορισμούς όπως ε, αναφέρεται από τον ΟΣΑ επίσης ένα σύστημα ε, επισημάνσεων που να διασφαλίζει το επίπεδο των, ε, των προϊόντων που παράγονται σύμφωνα με πρότυπα, πρότυπα περιβαλλοντικά για παράδειγμα την πρωτοβουλία που έλαβε σήμερα η Ιταλία σε ό,τι αφορά την επισήμανση στην καταγωγή των τομάτων που παράγονται με υπεύθυνο τρόπο. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, την πολυμερή προσέγγιση κλπ. Αυτή η έκθεση είναι καρπός πολλών ε, διαπραγματεύσεων για το πώς να χειριστούμε αυτή την παγκοσμιοποίηση. Έχουμε βρει ε, μια χρυσή τομή στην αναζήτηση ενός κοινού στόχου, δηλαδή για να γίνει ε, το εμπόριο ένα εργαλείο χειραφέτησης. Ένας συνάδελφος αναφέρθηκε στα σφάλω για τη Σιμόνε που έλεγε συζήτηση συμβιβασμού θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια λύση πιο ε, δυνατή που ε, παρά την θέση του καθενός. Αυτή η έκθεση καταδεικνύει αυτή την αναζήτηση. Ευχαριστώ τους ισχυώδεις συζητητές, ιδιαίτερα τον κύριο Ρώας που είναι σήμερα εδώ, που βρήκαν πραγματικά τους συμβιβασμούς που θα μπορούσαν να μας ικανοποιήσουν όλους και, και ελπίζω πολύ να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε. Και ξεκινούμε το KGI με τον κύριο Κέλλη. Ακούσα πολύ προσεκτικά ότι υπήρχε συγγήτρια. Νομίζω ότι γενικά ήταν πολύ ισορροπημένη η συνεισφορά της. Ως μέλος της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ Ξέρετε ότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το εμπόριο. Το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φυσικά αν παράγει αγαθά πρέπει να τα πουλήσει και φυσικά ω Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνάπτει εμπορικέ συμφωνίε που να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία όλων των κρατών μελών η συμφωνία ε, ε, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί αύξησε τις εξαγωγές κατά 50% ε, για τέσσερα χρόνια. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η λύση είναι να έχουμε εμπορικέ συμφωνίες αλλά να δούμε ε, ποια είναι τα αρνητικά και να διαβουλευτούμε με τα ενδιαφέροντα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι οι αρνητικές επιτυχίες ελαχιστοποιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καπούτα, ευχαριστώ. Η εμπορική πολιτική της Ένωσης, ε, κυρίως ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο, έχει γίνει μία από τις μεγάλες ε, ανησυχίες της κοινή γνώμας. Ε, συμφωνίες όπως η ΣΕΤΑ δεν μπορούν να επιβάλλουν μία εμπορική πολιτική. Διαμαρτυρίες που είδαμε σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύουν ότι οι ΜΜΕ αποτελούν το κεντρικό σημείο της παγκόσμιας αλυσίδα αξίας οι συμφωνίες ελεύθερων ε, συναλλαγών ε, ε, πνίγουν τους μικρούς παραγωγούς καθώς τους βάζουν να ανταγωνιστούν με επιχειρήσεις που δεν σέβονται τα ίδια πρότυπα ποιότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορική της πολιτική θα πρέπει να μείνει πιστή σε κάποιες αρχές και να καταπολεμήσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάπινγκ, να καταπολεμήσει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσει τις ιδιαιτερότητές της και τα σημεία που αριστεύει δεν μπορεί να συνεχίσει να τα ξεπουλά όλα αυτά μόλις είναι δυνατό. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών επί της ουσίας διάλυσαν τις οικονομίες των αναπτυγμένων κρατών και ταυτόχρονα άνοιξαν αγορές όπου εκεί επικράτησε η εκμετάλλευση των λαών για ένα κομμάτι ψωμί από τις πολυεθνικές και αυτό είναι ξεκάθαρο και αντιληπτό. ήρθε η ώρα λοιπόν να ληφθούν μέτρα και επομένως πρέπει να έχουμε σημαντικές πιέσεις στις χώρες όπου παράγονται τα προϊόντα από τις πολυεθνικές προκειμένου πρώτα απ' όλα να τηρούν την εργατική νομοθεσία να έχουν προσχωρήσει στις συμβάσεις της διεθνούς οργάνωσης εργασίας. δεύτερον θα πρέπει να υπάρξει ρήτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιπλέον πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε την παιδική εργασία και την εκμετάλλευση και την αναγκαστική εργασία. νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με το διεθνές εμπόριο. ευχαριστώ htio bih prije svega čestitati izvjestiteljici gospođi Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Αρένα για την εξαιρετική αυτή ε, έκθεση. Πρέπει να είμαστε νομίζω ανοιχτοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ηθικό ανάστημα για να δημιουργήσει τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα σήμερα στην συζήτηση και αύριο στην ψηφοφορία. Θέλω να τονίσω τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον είναι η εκμετάλλευση σε πολλές χώρες της φτηνής εργασίας, της υπερβολικά φτηνής εργασίας. Θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής ε, και της φορολογικής απάτης γενικώ ε, και της καταστροφής του περιβάλλοντος σε κάποιες χώρες. Είναι αυτό κάτι το οποίο τελικά πληρώνουμε εμείς, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ε, και βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες έχει συμφωνίες ελευθερού εμπορίου. Θεωρώ λοιπόν πως έχουμε μια συνολική έκθεση ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρένα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομο το ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικά μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο, την Επιτροπή Ίντα και την εισηγήτρια για τον χρόνο που επενδύσανε σε αυτή την έκθεση. Η Επιτροπή με το Ευρωκοινοβούλιο έχει κοινούς στόχους για την ατζέντα του 2030 για τις πολιτικές, ενλαμβανομένων των ε, πολιτικών εμπορίου και επενδύσεων η ε, εταιρική ευθύνη και όλα αυτά ε, υλοποιούνται από τους ε, εμπλεκόμενους μέσα από κανονιστικά μέτρα. Θα ήθελα να πω ότι η εταιρική ευθύνη είναι μια εθελούσια διαδικασία και έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ σε τις δράσει που έχουμε αναλάβει στον τομέα των παγκοσμίων αλυσίδων αξιών. Σε ό,τι αφορά την πολιτική αυτή, οι πρόσφατες ε, συμφωνίε ε, περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση τη βιομηχανία της ΠΑΑ. Η, η Κομισιόν προωθεί μέτρα στον τομέα των δημοσίων προμήθειών. Έχουμε εργαλεία κατά των πρακτικών διαφθοράς. Ε, και αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης ε, διατάξεις για την ε, εταιρική ευθύνη μαζί με άλλες, άλλα μέτρα για κοινά πρότυπα για περιβαλλοντικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται. Συνεργαζόμαστε με τον ΩΣΑ για να καταρτήσουμε έναν οδηγό για δέουσα επιμέλεια για την εταιρική ευθύνη μέσα από τον διάλογο στην, στα πρότυπα εργασίας και τις περιβαλλοντικές συμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα η Κομισιόν έχει ε, περαιτέρω πολιτικές ε, θα γίνουν περισσότερα ε, στην προώθηση της ενσωμάτωσης των ισότητας φύλων και επίσης σε ό,τι αφορά την ε, διάσκεψη του ΠΟΕ το 2017 σε ό,τι φορά τι άλλε πολιτικέ. Η Κομισιόν λαμβάνει μέτρα για τι παγκόσμιε αλυσίδε ε, αξιών. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτιση ε, δυνατοτήτων για να προωθηθούν μεταρρυθμίσει στον τομέα τη βελτίωση των προτύπων των εργασία και περιβαλλοντικών προτύπων. Επίση, βοηθάει τι μικρέ και μικρο, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με ε, την ΔΟΕ ε, στην βελτίωση των ε, συνθήκων εργασίας της Παγκόσμιας Αλυσίδας αξιών, επίσης και στο θέμα του κοινωνικού διαλόγου της εργασίας των παιδιών, καταναγκαστικής εργασίας. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες δικαιοδοσίας, συνεργαζόμαστε και διαπραγματευόμαστε μία σύμβαση ε, για ε, τη δικαιοδοσία με τρίτα μέλη. Επίσης έχει νομοθεσία για την εταιρική σχέση και την ε, υπεύθυνη συμπεριφορά των εταιριών. Υπάρχουν Υπάρχει μια οδηγία που απαιτεί από εταιρείε πάνω, από, πάνω από 500 ε, εργαζόμενους να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, διαφθορά κλπ. Και επίσης η οδηγία κατά της, του ξεπλήματος ε, υποχρεώνει επαγγελματίες να επιδεικνύουν διαφάνεια. Ε, αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα και πολλά άλλα θέματα και συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.